Good evening, colleagues. Uh, we will start. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε με τη συνεδρία της Επιτροπής. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα κάνουμε μια συζήτηση με την Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, την οποία ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ώστε να θέσουμε τα θέματα αυτά που ενδιαφέρουν ε, την Επιτροπή μας και θεωρούμε ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Για να οργανώσουμε λίγο τη συζήτηση θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Γιούροβα η οποία θα έχει χρόνο ε, γύρω στο 1 τέταρτο για να παρέμβει. Μετά θα ξεκινήσει ένας γύρος παρεμβάσεων. Θα ακούσουμε τους συντονιστές ή ε, εκπροσώπους των διαφορών πολιτικών ομάδων. Μετά θα μπορέσει να απαντήσει η κυρία Γιούροβα σε αυτά και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο συζήτησης για τους υπόλοιπους βουλευτές. Θα υπάρχει χρόνος παρέμβασης ώστε να μπορέσουν να λάβουν το λόγο όλοι. Στον πρώτο γύρο παρεμβάσεων λοιπόν θα έχουμε περίπου τρία λεπτά για τον καθένα για τους ε, ομιλητές ε, των πολιτικών ομάδων και στο δεύτερο γύρο παρεμβάσεων γύρω στο ένα λεπτό. Θα μπορούσα βέβαια να δείξω ευελιξία εάν δούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ε, παρατείνουμε λίγο τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Γιούροβα και να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσω μαζί σας σήμερα θέματα ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προτεραιότητες που πρέπει να ε, ε, εντοπίσουμε στον τομέα αυτό. Καταρχάς, ε, να δούμε λίγο την πολύ συντονισμένη και επιτυχή συμμετοχή στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των γυναικών το Μάρτιο στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι ειδικά το κοινό μήνυμα το οποίο αποστήλατε εσείς ε, και οι εκπρόσωποι ε, που είχατε στείλει, ήταν η πρόεδρος εκεί και κάποια άλλα μέλη, ε, εκπρόσωποι των κρατών μελών ε, και υποφαινόμενοι και τονίσαμε τη σημασία της ε, συνθήκης της Κωνσταντινούπολης και της αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Και ήμουν ιδιαίτερα περήφανη για μας ως ομάδα για την Ευρώπη, Team Europe, που ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα σαφές, ξεκάθαρο μήνυμα. Επίσης, ε, στα Ηνωμένα Έθνη είναι όλο ένα και πιο σημαντικό το θέμα αυτό, διότι πλέον η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να σταθώ στην ετήσια έκθεση για την ισότητα των φύλων που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο, η οποία επιβεβαίωσε ότι ακόμα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις προκειμένου η ισότητα των φύλων να υλοποιηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει φτάσει σε ένα ε, ε, ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο του 2015 εξακολουθεί να είναι 12% χαμηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Επίσης, το χάσμα το μισθοδοτικό εξακολουθεί να είναι αρκετά σημαντικό, όπως είναι και το χάσμα των συντάξεων. Ε, ούτε το μισθοδοτικό, ούτε το συνταξιοδοτικό χάσμα δεν ε, δείχνουν ότι θα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης. Υπάρχει ποσοστό προόδου στην ε, γυναική εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια. Ε, έχει βελτιωθεί στα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μέτρια αποτελέσματα. Το ένα τέταρτο και λιγότερο των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναικών και επομένως ε, πόρο απέχουμε ακόμα από την επίτευξη της ισότητας. Είναι ανησυχητικά επίσης ε, τα ποσοστά ε, της βίας. 33% των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή άλλη μορφή βίας. Και επίσης υπάρχουν και αρκετές εκκρεμότητες τις οποίες εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην ισορροπία ζωή ε, ζωής ε, και κουβίου. Ε, Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό και έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο. Έχουμε ε, μια διαδικασία αξιολόγησης των απαντήσεων που λάβαμε από τη δημόσια διαβούλευση και από την αρχική ανέλωση βλέπουμε ότι το μεγάλο ποσοστό των οργανώσεων, 97,8% καθώς επίσης και μεμονωμένα άτομα συμφωνούν με την περιγραφή των προκλήσεων που περιγράφουμε στο σχετικό έγγραφο. Το 85% συμφωνεί ότι ο κατάλογος ε, των τομέων πολιτικής στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ο σωστός κατάλογος. Οι τομείς πολιτικής είναι η φροντίδα των παιδιών, μακροχρόνιες υπηρεσίες φροντίδες, ε, άδεια ε, για την οικογένεια, οικογενειακή άδεια και για άνδρες και γυναίκες, ε, ευέλικτο ωράριο εργασίας και για άνδρες και γυναίκες, ε, φορολογικά κίνητρα και για τους δύο γονείς ώστε ε, να εργάζονται. Το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους θα ξεκινήσει σύντομα και η Επίτροπος και, Τάισεν και εγώ θα σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά μέσω επιστολής. Εάν οι κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν να μην διαπραγματευτούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόθεση να προτείνει μια δέσμη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που θα αντιμετωπίζουν ε, τις διάφορες πτυχές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις ε, για το γεγονός ότι μόνο έξι κράτη-μέλη έχουν επιτύχει τους στόχους της Βαρκελόνης για ε, εγκαταστάσεις για ε, την ε, μέρημνα των παιδιών και επίσης τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ε, σημερινή εργασιακή πραγματικότητα, κυρίως ε, τα πλεονεκτήματα της, ψηφιακής, της ψηφιακής εποχής για ευέλικτα ωράρια εργασίας και τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι περισσότεροι άνδρες θα ήθελαν να αναλάβουν περισσότερες ε, αρμοδιότητες και καθήκοντα για τη φροντίδα των παιδιών του στην οικογένειά τους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί προς αυτό. Ευπρόσδεκτο το εύρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως τη Επιτροπή Γυναικών και Απασχόλησης, για πρωτοβουλία για την ισορροπία εργασιακού ε, βίου και ε, ε, οικογενειακής ζωής και επίσης το γεγονός ότι θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να συνεργάζεστε μαζί μας ως σημαντικός εταίρος σε αυτή τη σημαντική προπαρασκευαστική διαδικασία και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι θα υπάρχουν και συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξωμήνου όπου αναμένεται οι ελλείψεις για την συμμετοχή των γυναικών ε, στην ε, εργατική ζωή να αντικατοπτρίζονται με κάποιο τρόπο. Επίσης, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το χάσμα ε, στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή του και τι συνέπειες υπάρχουν για τα κράτη-μέλη και θα έχουμε και κάποια επόμενα βήματα για ενισχυμένα νομοθετικά μέτρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης ε, και οι οποίες συνεχίζονται και υπάρχει και συνεργασία με τους φορείς ισότητας ε, που διευκολύνουν την εφαρμογή της αρχής της ίσης ε, ε, αμοιβή για την αντίστοιχη εργασία στα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, στο θεματολόγιο για τις ε, δεξιότητε και τα επαγγελματικά προσόντα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον εργασιακό διαχωρισμό ως μία από τις ρίζες του χάσματος που υπάρχει μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών. Να σας... πω δύο λόγια για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος των γυναικών. Όπως σας επισημάνθηκε και αναφέρθηκε προηγούμενα κατά το παρελθόν, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είμαι πεισμένη ότι αυτή η προσχώρηση μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά για τις ζωές κοριτσιών και γυναικών, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβουν βήματα και διαβήματα για να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα της βίας εις βάρος των γυναικών και θα συνεργαστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει παράλληλα με τα κράτη-μέλη, δεν θα υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη. Σημαντικές πτυχές αυτής της σύμβασης που όσον αφορά τα θέματα τα νομοθετικά θα παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και έτσι θα έχουμε πρόσθετα ωφέλη από αυτή την προσέγγιση την ευρωπαϊκή. Θα έχουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές, καλύτερη χρήση κονδυλίων, βελτιωμένη συλλογή δεδομένων και θα έχουμε αξιόπιστη φωνή που θα αρθρώνουμε με τους ε, ε, οικουμενικούς εταίρους μας. Η απόφαση από πλευράς ε, θα απαιτήσει τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε έτσι. Και ευελπιστώ ότι η κοινοβουλευτική σας επιτροπή θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποστείλει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη για αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Για να καταπολεμηθεί η βία εις βάρος των γυναικών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και η νομοθεσία, η συλλογή στοιχείων και η χρηματοοικονομική υποστήριξη για πρωτοβουλίες επιτόπου, ευαισθησία και ευαισθητοποίηση. Διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Μόνο αλλάζοντας νοοτροπίες και συμπεριφορές μπορούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τη βία εις βάρος των γυναικών προτού εκραγεί διασφαλίζοντας ότι θα καταδηλώνονται, θα αναφέρονται στις αρχές ε, αυτά τα περιστατικά και τα θύματα θα την χάνουν σημαντική ευαίσθητης υποστήριξης όπως δικαιούνται. Εγώ έχω υπόψη να προχωρήσω στοχοθετημένες δράσεις ε, υπέρ των γυναικών που αποτελούν ε, στόχους αυτής της βίας. Προβληματιζόμαστε και σκεφτόμαστε για το εύρος ε, και την κλίμακα αυτών των δράσεων για να έχουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για αυτές τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε χρήση όλων των εργαλείων και μέσων στη διάθεσή μας. Δηλαδή ευαισθητοποίησης ε, με κάθε τρόπο να υποστηριχθούν ε, οι πολίτες ε, στη βάση τους και τα κράτη-μέλη για τα πρότυπα όσον αφορά τα, τα θύματα και τις αρχές που πρέπει να είναι σεβαστές πάντα και θα ανταλλάξουμε και βέλτιστες πρακτικές και προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να γίνουν όλα αυτά. Επίσης θα ενημερώνω σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν θα υπάρχει ενημέρωση όσον αφορά τα θύματα, όπως και την εντολή προστασίας των θυμάτων, ευρωπαϊκή εντολή, καθώς επίσης και την υποστήριξη ε, μέσω δράσεων που θα καταπολεμούν την ανθρωποεμπορία και θα υποστηρίζουν τα θύματα. Συλλογή δεδομένων ως απαραίτητη βάση για αυτές τις μελλοντικέ προσπάθειές μας. Χαίρομαι που έχουμε την επιβεβαίωση, την επαλήθευση από την Ευρωστάτ ότι θα αρχίσουν εργασίες εφέτος για τη συλλογή δεδομένων για την, τα θέματα βίας εις βάρος των γυναικών. Ένα άλλο σημείο κλειδί ως πεδίο σε αυτή τη μάχη είναι να υπάρξει η καλύτερη ισορροπία όσον αφορά θέματα φύλων στις λήψεις αποφάσεων. Η συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι στόχος μας ως δεσμευτικό μέσο ώστε να υπάρξει πάγια και ισχυρή πρόοδος που θα σημειωθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι εδώ μεγαλύτερη προσπάθεια και πρόοδος έχει, έχει σημειωθεί στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εξέταση νομοθετικών δράσεων. Βλέπουμε ότι αυτά τα νομοθετικά μέτρα οδηγούν σε αποτελέσματα. Μία πλειοψηφία των κρατών μελών υποστηρίζει την προτινόμενη οδηγία. Θλίβομαι για το ότι κάποια κράτη δεν δείχνουν ακόμα την ε, όριμη πολιτική βούληση που απαιτείται στο πολιτικό επίπεδο υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Καλωσορίζω την απόφαση όσον αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου να αποτελέσει προτεραιότητα αυτή η δράση και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ως Επιτροπή την προσπάθεια να επιτευχθεί αυτό το, η θετική έκβαση με σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο να ασκηθεί πίεση για τις τρέχουσες εργασίες ε, όσον αφορά την τρέχουσα Προεδρία αλλά και τις μελλοντικές Προεδρίες ώστε να υπάρξει υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όπως όλοι γνωρίζουμε την χρειαζόμαστε πράγματι κατεπηγόντως επιτακτικά. Να αναφερθώ τώρα στο θέμα της μετανάστευσης και της ε, κατάστασης ε, των μεταναστριών γυναικών. Σίγουρα πρέπει η ένταξη του φύλου στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις δράσεις μας να ενταχθεί σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι ένα σύνθετο και περίπλοκο θέμα και απαιτεί βραχυπρόθεσμα άμεσα μέτρα όσον αφορά για παράδειγμα τα hot spots και την υποδοχή, αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και παιδεία. Γνωρίζω ότι έχετε αρθρώσει λόγο και φωνή από αυτών των θεμάτων και προσβλέπω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε συνεργαστούμε ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας. Θα συζητήσουμε και τα θέματα αυτά με τους υπουργούς των κρατών μελών που εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να υπάρξει αυτή η συμμετοχή. Στο τέλος συνεργαζόμαστε στενά όσον αφορά το Ίδρυμα για την ισότητα γυναικών και ανδρών. Θα συνεχίσει το Ίδρυμα αυτό να παρέχει πλαίσια για τις πολιτικές μας εφέτος από πλευρά ΕΓΕ του ιδρύματο για την Ισότητα των Φύλων θα υπάρξει μια έκθεση όσον αφορά την φτώχεια των γυναικών για παράδειγμα και την κατάσταση των γυναικών και προσβλέπουμε στο να ενταχθούν αυτά τα θέματα σε σχέση με τους δείκτε το 2017. Για πρώτη φορά θα συλλέγονται έτσι στοιχεία όσον αφορά την ε, ε, επίδραση, την επίπτωση που έχει η ε, άνηση μεταχείριση και οι ανισότητες εις βάρος των γυναικών. Θα υπάρξει έτσι λοιπόν και εξέταση των ε, δράσεων για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ για την επικοδομητική σας υποστήριξη στις προσπάθειές μου μέχρι σήμερα να καταλήξουμε σε χειροπιαστά συγκεκριμένα αποτελέσματα για την ισότητα των γυναικών. Και προσβλέπω και περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιουροβά για την παρουσίασή σας. Ξεκινάμε με τις παρεμβάσεις των ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, η κυρία Λεγκρίπ, η κυρία Λεγκρίπ παρακαλώ, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για την παρουσίασή της αλλά και για την ε, συνεχή διαθεσιμότητά τη. Είναι πάντα διατεθειμένη να έρθει εδώ, να μιλήσει ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Είχαμε πολλές ευκαιρίε ε, να διαπιστώσουμε και τη δική σα ε, ε, προσωπική αφοσίωση σε αυτό το ζήτημα το οποίο και εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Για τα επιμέρους ζητήματα που θίξατε, εγώ θα σταθώ σε ένα και η Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ συντονίστρια του ΕΛΚ θα μπορέσει να πάρει το λόγο στη συνέχεια για να αναφερθούμε από κοινού στα ζητήματα που αφορούν για μας προτεραιότητες. Βεβαίως δεν είναι κλειστός αυτός ο κατάλογος θεμάτων. Μιλήσατε για το μισθοδοτικό και σταξιδιωτικό χάσμα. Και πολύ σωστά είπατε ότι δεν μειώνονται και τόσο πολύ αυτά τα χάσματα. Παραμένει λοιπόν αυτό το χάσμα και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και τους συμπολίτε μας, ιδίως με τη γύρα του πληθυσμού. Πλέον αυτό το θέμα λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πιο σημαντικό. Το είδαμε και με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε και με τα συμπεράσματα των Ιούνιο του 2015. Ε, είδαμε ότι έχει δοθεί έμφαση σε αυτά τα ζητήματα. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πλέον χρήσιμο μέσο για εργαλείο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για να δώσουμε ένα τέλος και επιτέλους να καταφέρουμε να κινήσουμε τα κράτη-μέλη προς ε, τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται μία ομοιόμορφη προσέγγιση, αλλά ε, πιο ευέλικτα και κλεπτισμένα εργαλεία, τα οποία θα ήταν πιο κατάλληλα. Ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που εσείς ε, θα επιλέξετε στους επόμενους μήνες και δύο λόγια για το Women on Boards, τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Εμεί βεβαίω ε, συμμετέχουμε στι πολιτικέ δυνάμει που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, τους, ώστε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν τη σημασία προώθησης αυτού του σημαντικού φακέλου. Παρότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτή τη διαδρομή μαζί σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέτ, ε, παρακαλώ, των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θα θέλουν να ευχαριστήσουν την κυρία Γιούροβα για τη δυνατότητα ε, που μας δίνει να την ακούσουμε σήμερα και να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα μαζί της στην Επιτροπή Γυναικών. Για τους ε, στόχους ε, της Βαρκελόνης, εγώ είμαι εδώ αρκετά χρόνια πλέον και δυστυχώς βλέπουμε ότι πολύ λίγα κράτη-μέλη έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αναλάβουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε να δίνεται δυνατότητα αγωνικής άδειας σε όλους καθώ και σε ό,τι αφορά την παιδική μέρημνα που θα βοηθήσει και τι γυναίκε να επανέλθουν στην αγορά εργασία. Όμω και εσεί είπατε ότι δεν έχουν γίνει ε, όλα τα δυνατά για να αρθούν αυτά τα προσκόμματα. Επίσης, Λυπάμαι που η στρατηγική έχει αποδυναμωθεί από νομικής ε, άποψης. Θεωρώ ότι στα κράτη-μέλη ε, θα μπορούσαν να έχουν ανατεθεί μεγαλύτερες αρμοδιότητες για να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια. Επομένω, η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, θεωρεί λυπηρό ότι δεν υπάρχει μία εύρωστη στρατηγική. Από οικονομική σκοπιά, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία ήταν επωφελή προ όλου και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για να προωθήσουμε αυτό το μέτρο. Τώρα για την οδηγία για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Women on Boards. Είπατε ότι έχετε λάβει βήματα ε, για αυτό το ζήτημα, όμως διερωτώ τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Μετά έχουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία Ούτω ώστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο θεσμικών οργάνων, θα υλοποιήσουμε την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε πολλά. Είναι κρίμα βέβαια που δεν συμπεριλαμβάνονται και αυτά τα ε, δικαιώματα, γιατί ξέρουμε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχουν ποινικέ κυρώσει για τη βία κατά των γυναικών, όμω χαίρομαι που ελήφθη αυτή η απόφαση. Ευχαριστώ κυρία Μιλνάρ από την ΑΛΔΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο που είναι εδώ μαζί μας και για την ανταλλαγή απόψεων για όλα αυτά τα κέρια ζητήματα που παρουσιάσατε. Το εκτιμούμε και από πλευρά ε, φιλελευθέρων. Ορισμένα ζητήματα που και εσεί στήξατε, αλλά θα θέλω να τα αναφέρω και εγώ, γιατί ήμασταν όλοι μαζί στη Νέα Υόρκη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει για πρώτη φορά ε, τόσο προβλημένο ρόλο και ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ρόλο στα επόμενα χρόνια, αλλά ήταν καλό βήμα. Τώρα, σε αφορά τα συμπεράσματα για την κατάσταση των γυναικών. Είναι μακρόπνοα βεβαίως ε, και ως ήθη στις τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων. Όμως, ποιες είναι οι δικές σας απόψεις Ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων ω προ την ισότητα των φύλων. Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα ευρύ το θέμα, αλλά είχαμε όλοι νομίζω την εντύπωση ότι ήταν ε, ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή η συνάντηση. Επομένω, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δική σα άποψη για τον ρόλο μα στο διεθνέ προσκήνιο. Δεύτερον, Κάτι το οποίο αναφέρατε, επίσης αναφέρατε. Για τις ε, γυναίκες ετούντες άσυλο και το πόσο ευάλωτος είναι. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε και στο Σώμα των Επιτρόπων. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει και δεν πρόκειται να φύγει με στου επόμενου μήνε ή ακόμα και χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα προληπτικά μέτρα και όσο προ αυτό. Και τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της στρατηγικής ισότητας των φύλων. Να μας πείτε με δύο λόγια κάτι γι' αυτό. Και τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πιέσεις ε, που ασκείτε και στο Σώμα των Επιτρόπων για την ε, ε, προσχώρηση στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, γιατί δεν είναι μόνο ε, κάτι το τυπικό, είναι και ένα πολιτικό μήνυμα. Και γνωρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι και εσείς προσωπικά ε, το προσπαθείτε. Ευχαριστώ. E. Ευχαριστούμε εξ ονόματος της ΓΚΟΕ e, Άβια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ θερμά το ότι προσήλθατε εδώ στην Επιτροπή μας κυρία Γιούροβα και έχετε την προθυμία να συζητήσετε μαζί μας. Δεν θα σας εκπλήξει αν σας πω ότι από πλευράς της Ενωτικής Αριστεράς εξακολουθούμε να έχουμε την εντύπωση ότι στα θέματα ισότητας υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εκκρεμούν και ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί όταν ζητούμε να υπάρξουν γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, αυτό ο στόχος είναι ανεπαρκέστατος και η κατάσταση αυτή είναι ως έχει σήμερα πραγματικά παράδεκτη και οι προσπάθειες που καταβάλλονται πρέπει να μας κάνουν να αντιμετωπίσουμε και την βία εις βάρος των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό χρειάζονται αυτές οι δράσεις. Χαιρετίζουμε επίσης τις προτάσεις που εσείς ε, ε, υποβάλλατε για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα, οι μισθολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών. Η θέση των γυναικών στην εργατική ε, ζωή θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Καθώς επίσης και σε σχέση με την περίθαλψη των υπερηλίκων είναι σε μειονεκτική θέση οι γυναίκες, εξακολουθούν να είναι σε μειονεκτική θέση και πρέπει να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Προσβλέπουμε, αναμένουμε, αδειμονούμε να δούμε την πρότασή σα για τη γονεϊκή άδεια. Και εδώ, ναι, μεν συζητάμε για σημαντικά θέματα, όμως δεν μπορούμε να αμελήσουμε και να αγνοήσουμε ότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ακριβώς ποια είναι η συνολική θέση της Επιτροπής όσον αφορά τα θέματα ισότητας σφαιρικά. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πιέζουν διαρκώς ε, για αυτή την κατεύθυνση. Εσείς δεν έχετε καταλήξει σε μια τέτοια ενιαία στρατηγική. Αν υπάρχει μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να επιλεγούν συγκεκριμένες προτάσεις, ε, άλλες προτάσεις θα πρέπει να αφαιθούν στο περιθώριο, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει μια στρατηγική, ενιαία στρατηγική. Στρατηγική σημαίνει συμφωνία συμφωνία μεταξύ εταίρων. Έτσι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να είναι εταίροι, σύμμαχοι για να καταλήξουν προς μια ενιαία κατεύθυνση. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να προαγάγουμε τα θέματα ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθούν και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι επίσης σημαντικό να δούμε από την άλλη πλευρά την ενδυνάμωση των γυναικών σε θέσεις ε, που θα λαμβάνουν αποφάσεις οι γυναίκες. Όχι μόνο την ε, συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, δεν θέλουμε απλά μόνο κάποιες εκατοντάδες γυναίκες να ενταχθούν σε διοικητικά συμβούλια και μετά να πούμε ότι επακούμαστε με αυτό. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά να έχει μια σφαιρική θέση για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και για τους πράσινους η κυρία Ρέτκε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ από πλευρά μου να σας ευχαριστήσω που έχουμε μια σχεδόν μόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Χαίρομαι που έρχεστε τόσο τακτικά στην Επιτροπή και πιστεύω ότι από αυτά που ακούμε και από εσά, ε, η ανησυχία μα όσον αφορά την ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινέ. Γι' αυτό και θα είμαι και λίγο ομοί για τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την κατάσταση αυτή τη στιγμή και να σα πω και κάποια παραδείγματα και να εμβαθύνομαι λίγο στη συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Διότι αυτό που διαπιστώνω αυτή τη στιγμή ε, είναι ότι υπάρχει μια μειοψηφία που επιτίθεται στην ισότητα και στα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η αναστέλουσα μειοψηφία όχι μόνο δεν επιτρέπει να υπάρχει καμία πρόοδος, αλλά επιτίθεται και σε πάγιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να υπάρχει μια βαθύτερη στρατηγική για να το καταπολεμήσουμε αυτό. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι είχαμε ανταλλαγή απόψεων με την Ολλανδική Προεδρία σήμερα το πρωί και μία από τις προτεραιότητες ε, που έθεσαν ήταν ε, ο δικός χάρτης για τους ΛΟΑΔΜΑ. Και η Ουγγαρία δεν ήθελε να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και ξέρω ότι ο δικός χάρτης και η στρατηγική για τους ΛΟΑΔ αποτελεί και δική σας προτεραιότητα. Επομένως θεωρούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου είμαστε όλοι ενωμένοι για να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά και υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων στο Συμβούλιο που δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο πιαστικοί ώστε να υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτή την αναστολή των τόσο σημαντικών θεμάτων. Και αυτό δεν είναι μόνο για, την, ε, για τον οδικό χάρτη. Αναφερθήκαμε και για την, στην οριζόντια στρατηγική για την ισότητα, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τα θέματα εξισορρόπησης οικογενειακού και εργασιακού βίου και βλέπουμε ότι πάντα υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ε, αποτελούν τροχοπέδι στα θέματα αυτά και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να θίξω είναι το γεγονό ότι θα μάθετε ότι εγκρίθηκε έκθεση για την προώθηση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Δεν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό στην εισαγωγή σας, αλλά νομίζω ότι η επιρροή που μπορείτε να ασκήσετε εσείς ως Επίτροπος υπεύθυνη για την ισότητα των φέλων, για παράδειγμα σύγκληση για τις ψηφιακές ε, θέσεις εργασίας και το όλο ψηφιακό θεματολόγιο για να προθέσετε τη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των φύλων ε, σε σχέση με την ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον ε, σκοπεύετε, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα στη Μικρή Ολομέλεια θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση, θεωρώ ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συμμετοχή και σε αυτή τη συζήτηση, ώστε να έχουμε ένα θεματολόγιο το οποίο ασχολείται με όλα τα θέματα και που θέτει την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρέντε και τέλο, επειδή ολοκληρώθηκε ο πρώτο γύρος παρεμβάσεων των πολιτικών ομάδων, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιούροβα για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα διατρέξω όλες τις ερωτήσεις. Κάποιες βέβαια ερωτήθηκαν από πολλούς. Ε, κύρια Λε Γκρίπ, μισθοδοτικό χάσμα και συντάξεις. Συμφωνώ μαζί σας. Πού είναι, σας έχασα. Ήθελα να σας απαντήσω. Αλλά έφυγε η κυρία Λεγκρίπ. Για το θέμα αυτό πρέπει να είμαι ιδιαίτερα ανοιχτή μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε σπουδαία αποτελέσματα από την όλη διαδικασία διαφάνειας, διότι συλλέγαμε τα δεδομένα, με ε, προθεσμία το πέρας του προηγούμενου έτους, αλλά αυτή τη στιγμή τα αξιολογούμε. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε το χάσμα μισθών μόνο πιέζοντας ε, τη διαφάνεια, μόνο πιέζοντας τους εργοδότες να ενημερώνουν για την πολιτική ε, των μισθών που εφαρμόζουν. μπορεί να τους οδηγήσει στο να το σκεφτούμε, αλλά δεν νομίζω ότι ε, θα αλλάξει πολύ την κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις τρεις πηγές για το χάσμα μεταξύ των μισθών. Το ένα είναι ανοιχτή διάκριση. Ένας άνδρας μπορεί να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα για την ίδια θέση εργασίας. Εδώ αυτή είναι η σαφής ε, κατάσταση. Εδώ έχουμε την οδηγία για ίση μεταχείριση και κατά των διακρίσεων, η οποία ε, περιλαμβάνει κυρώσεις. Και δεν έχουν κατάλληλα μέσα όλα τα κράτη-μέλη για να επιβάλλουν κυρώσεις ε, όταν υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση, όταν άνδρας, ε, χωρίς να υπάρχει κανένα σοβαρός λόγος, πληρώνονται περισσότερο από τις γυναίκες. Σκοπεύουμε λοιπόν να προωθήσουμε την οδηγία και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα μέσα, ώστε οι εργοδότες να μην ε, ε, ε μένουν ατιμόρυτοι. Όμως, η διάκριση αυτή δημιουργεί μόνο ένα 8% των ε, προβλημάτων στο μισθό. Υπάρχουν διακρίσεις λόγω των θέσεων εργασία. Ξέρετε, για παράδειγμα, τι γίνεται με νοσοκόμες, ε, δασκάλους, και εδώ αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο αποτελεσματικό μέτρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από ευρωπαϊκή σκοπιά ώστε να υποχρεωθούν τα κρατημένα να αλλάξουν την πολιτική του. Θα ξανασυζητηθεί όμω το Συμβούλιο Έψικο του Ιουνίου, διότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ε, ε, όσον αφορά τις διαφορές της συντάξης, διότι είναι προβλήματα τα οποία αποδεικνύουν ότι αν δεν αλλάξει το σύστημα ε, ασφαλίσεων και κοινωνικών ε, ε, επιδομάτων δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό όμως είναι στα χέρια των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και με τη νέα δέσμη μέτρων για την ισορροπία οικογενειακού και εργασιακού δίου. Μπορεί να υπάρχει μια παγίδα εδώ και να εκμεταλλεύονται περισσότερο οι εργοδότες ε, τις θέσεις μερικές απασχόλησης, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μικρότερη μισθοδοσία, χαμηλότερους μισθούς. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει κάτι τέτοιο, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες και να κάνουν παιδιά και να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα για ευέλικτες μορφές εργασίας και να μπορούν φυσικά να εξοικονομούν και τα προστοζήν, ε, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και εμάς ε, να μειώσουμε το χάσμα αυτό μεταξύ μισθών. Ε, αν έχετε κάποιες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε για κάποιες ε, ε, θέσεις εργασίας που αποτελούν διάκριση, ε, ενημερώστε μας. Δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε ποσοστώσεις για τους άνδρες, σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επικρίσεις για τις ποσοστώσεις ήδη. Τώρα, η τρίτη πηγή για το χάσμα μεταξύ των μισθών, είναι χαμηλή αυτή η εκτίμηση των γυναικών και των κοριτσιών και φυσικά και τη, οι επιλογές που κάνουν ως προς την μόρφωσή τους. Οι γυναίκες σπουδάζουν σε τομείς που δεν πληρώνονται πάρα πολύ καλά και δεν έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε ώστε το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες, αν παρακολουθείτε τι κάνουμε στον τομέα της παιδείας και της ε, πολιτικής εργασίας, παρακαλώ εξετάστε το γιατί προσπάθησα πολύ σκληρά να εξονθρολογήσω και τα θέματα ισότητας των φύλων ε, και να τα εντάξω σε αυτήν την τόσο σημαντική νέα πολιτική, διότι πρέπει να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια ώστε να σπουδάσουν ε, κατάλληλα ε, επαγγέλματα, ώστε όπως λένε και οι επικεφαλείς επιχειρήσεων τεχνολογίας να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διότι όποτε συζητώ μαζί τους ε, πιέζω για καλύτερες πιθανότητες για τις γυναίκες να τους ε, θέσω σε μια θέση ε, να λαμβάνουν αποφάσεις και να λαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και συνεχώς μας λένε ότι δεν έχουμε στις γυναίκες στην πρώτη γραμμή γιατί δεν σπούδασαν το κατάλληλο αντικείμενο. Και νομίζω ότι αυτό εν μέρει αληθεύει. Εξακολουθούν να ισχύουν κάποια στερεότυπα, ιδίω σε επιχειρήσει τεχνολογία. Μου λένε ότι δεν υπάρχουν γυναίκε μηχανικοί και του λέω ότι ίσως θα μπορούσαν να πάνε εμπειρογνώμονες από τον τομέα του μάρκετινγκ και οι νομικούς συμβούλους ε, καταρχάς και εκεί σταματάει φυσικά η συζήτηση γιατί ε, υπάρχουν συγκεκριμένα στερεότυπα. Για τους στόχους της Βαρκελόνης, είναι εντυπωσιακό πόσο το θέμα της έλλειψης υποδομών ε, για την παιδική μέρηχνα ε, επηρεάζει πάρα πολύ τις διαβουλεύσεις μας για την ισορροπία οικογενειακού και εργασιακού βίου. Ε, εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκες ή μάλλον οι ίδιοι οι γονείς χρειάζονται κατάλληλες υποδομές για να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους ώστε να πάνε ε, να εργαστούν. Αλλά υπάρχει έλλειψη τέτοιων υποδομών σε πολλά κράτη-μέλη και πραγματικά εγώ ενθαρρύνω ε, τους ε, αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με κάποια μορφή κονδυλίων για επενδύσεις, να αλλάξουν οι προτεραιότητες για τα κράτη-μέλη, διότι φέτος είναι η χρονιά της αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα κράτη-μέλη τα οποία ε, θα θέσουν νέες προτεραιότητες θα μπορούσαν ίσως να προτείνουν και αλλαγές. Αυτό είναι εξελίξη. Δεν ξέρω πόσα κράτη-μέλη θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι και θέμα χρημάτων. Επίσης, ε, εδώ υπησέρχονται και τα στερεότυπα. Γυναίκες οι οποίες θέλουν να μείνουν περισσότερο με τα παιδιά τους, ε, υποτίθεται και δεν θέλουν να τα στείλουν ε, σε ένα βρεφιονιπιακό σταθμό και παιδικό σταθμό πριν τα παιδιά κλείσουν τα τρία χρόνια. Αλλά υπάρχει και κάτι καινούριο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία για την ε, πολιτική ένταξη ε, των Ρωμά διότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ήδη διαθέτουν σχετική νομοθεσία και προβλέπουν τα παιδιά των Ρωμά από την ηλικία των 4 ή 5 ετών να ε, πηγαίνουν υποχρεωτικά στον υπηαγωγείο ώστε να προετοιμάζονται για το δημοτικό. Αυτή είναι άλλη ιστορία βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα το θίξω κάπου αλλού. Τώρα, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια τώρα, πού βρισκόμαστε. Ε, κάποιοι είπατε ότι χαίρεστε που βρισκομαστε καποιοι ειπατε οτι τακτικά και χαίρομαι που σας ακούω να το λέτε αυτό, αλλά κάθε φορά σκέφτομαι τι καινούριο μπορώ να σας πω. Για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβόλαια δεν έχω και πολλά να σας πω περί πρόοδου, γιατί είμαστε εκεί που βρισκόμασταν και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει. Εξακολουθούμε να περιμένουμε δύο από τα μικρότερα κρατημέλη και ένα από τα μεγαλύτερα να ε, σταματήσουν την αναστέλουσα μειοψηφία ε, στο Συμβούλιο Εξακολουθούμε να είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία, τις κάτω χώρες και τη Δανία, την Ουγγαρία επίσης. Άλλος κανείς ή κάτω χώρες της Ήπα, τις κάτω χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε να αλλάξουμε στη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας του χρόνου. Εν τω μεταξύ, σας υποσχέθηκα εδώ ότι θα συνεργαστούμε στενά με τις ίδιες τις επιχειρήσεις και αυτό κάνουμε. Είμαι σε πολύ συχνή επαφή με τις ε, ε, εισηγμένες ε, εταιρείε και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι για αυτούς είναι καλύτερα να το ξεκινήσουν επί εθελοντικής βάσεως και να μην τους υποχρεώσουν νομοθεσία να το εφαρμόσουν. Αλλά, εντάξει, αυτό το λέω αστευόμενοι μεν, αλλά οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ε, ότι η ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια είναι καλή και είναι χρήσιμη για τις επιχειρήσεις τους. Και πολλοί από αυτούς έχουν εσωτερική επιχειρηματική στρατηγικές και στρατηγικές περί ανθρωπίνων πόρων και θέλουν να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι σταδιακά, ακόμα και χωρίς νομοθεσία, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο, αλλά με νομοθεσία την οποία ε, θα προσπαθήσουμε να ε, ε, περάσουμε, θα έχουμε ίσως πρόοδο νωρίτερα. Για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ναι, πράγματι, θέλουμε να εγκριθεί φέτος σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε τρία κράτη-μέλη, τα οποία ακόμα δεν έχουν κυρώσει νομίζω. και 15 που δεν έχουν ούτε υπογράψει ούτε κυρώσει. Αλλά πιέζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης οδηγεί σε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Και μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα από αυτόν. Επομένως πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Πρόκειται περί μεικτής συμφωνίας και πρέπει να κάνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και εγώ θεωρώ ότι είναι και μια πρακτική ε, πράξη νομοθετική και εδώ ε, φτάνω και στο θέμα της βίας και θα ήθελα να σταθώ λίγο εδώ στη βία γιατί θα ήθελα να σας ζητήσω για ιδέες για το 2017. Το 2017 θέλουμε να το ανακηρύξουμε έτος καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και θέλουμε να γίνει και με τρόπο που θα μας οδηγήσει σε αποτελέσματα. Να είναι ένα συνδυασμό μιας εκστρατείας που θα είναι μια γενική εκστρατεία σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Ε, δεν θα υπάρχουν πολλά σε αυτή την πανευρωπαϊκή εκστρατεία γιατί είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών δεν πρέπει ε, το ξυπνητήρι μου ήταν αυτό που χτύπησε. Ε, πλάκα κάνω. Στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές μορφές ε, βίας και με διαφορετική ένταση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχει θέμα οικογενειακής βίας. Στη Γερμανία πλέον διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν περιστατικά βίας σε δημόσιους χώρους. Ε, υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα γιατί η βία εμφανίζεται στις ε, εθνικές μειονότητες. Επομένως πρέπει να υπάρχουν στοχευμένες εκστρατείες ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία διαπιστώνουμε σε κάθε κρατός μέλος. Γι' αυτό και χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα από τους υπουργούς στη Νέα Υόρκη, γιατί ε, συναντήθηκα με τους ε, υπουργού κατά την σύνοδο στη Νέα Υόρκη υπεύθυνου για θέματα ισότητας των φύλων, ότι σκοπεύουν να συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη δράση για το 2017. Θα ε, τους στείλω επιστολή την επόμενη εβδομάδα, διότι ήθελαν να τους ε, δώσουμε ιδέες για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε και φυσικά υπάρχει ένας πρακτικός λόγος, θέλουν να το εντάξουν και στον προϋπολογισμό τους για το 2017. Πραγματικά λοιπόν ε, το εννοούν. Όταν ένας υπουργός λέει ότι θα το συμπεριλάβω στον προϋπολογισμό μου, σημαίνει ότι εννοούν ότι θα κάνουν κάτι από αυτού. Αυτή θα είναι η κοινή μας δράση. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και συγχρηματοδότηση ε, των εξτρατιών των κρατών μελών, αλλά θα υπάρχει και ένα ε, σημείο εξορθολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει στρατηγική δεν αφορά το θέμα όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ε, υπήρξαν πολύ θετικές αντιδράσεις από τον συνάδελφο Ναυράτσης, Ανδρουκάητης, ε, για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλεια και του απίθυνα και έκκληση ε, να μας προτείνουν κάποιες ιδέες για το πώς θα συμμετέχουν και οι ίδιοι στην εκστρατεία. Θα χρηματοδοτήσουμε και τις ε, βασικές οργανώσεις, μη κυβερνητικούς και οργανώσεις, θα εκπαιδεύσουμε και εμπειρογνώμονες και θα ήθελα εδώ να μου πείτε κι εσείς κάποια πράγματα για το κατά πόσο θεωρείτε ότι σκεφτόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση θεωρώ ότι πρέπει να αποτανθούμε και στις γυναίκες και στις αρχές επιβολής του νόμου, δηλαδή αστυνομία, ε, δημοτική αστυνομία που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των πολιτών. Ε, και αυτό, ε, γιατί αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Οι γυναίκες δεν κάνουν καταγγελίες γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τους βοηθήσει και κανείς. Επίσης πρέπει να αποφθυνθούμε και στους άνδρες και στα αγόρια, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο μείγμα για την εκστρατεία και πραγματικά να στοχεύσουμε στις σωστές ομάδες. Αυτά λοιπόν περί βίας. Θα σας στείλω σχετική επιστολή λοιπόν και θα ζητήσω τις προτάσεις σας. Η κυρία Μπιόρκ για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Κύριε Μάρκετα, τα δύσκολα ερωτήματα που έθεσε. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διεθνές ε, πλαίσιο και τις διεθνείς επαφές. Στη Νέα Υόρκη, βεβαίως επικεντρωθήκαμε κυρίως στα ευρωπαϊκά ζητήματα, ιδίως αυτό της ε, μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστριών. Όμως, ό,τι αφορά τις ε, εξωτερικές δράσεις, υιοθετήσαμε μια δέσμη μέτρων ε, με γνώμονα τη διάσταση του φύλου, με συγκεκριμένους δίκτες, κυρίως ό,τι αφορά την ε, ακαιρεότητα και αξιοπρέπεια των γυναικών. Και αυτό μας ξαναφέρνει στις προσπάθειες εξάλληψης ε, της βίας κατά των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο αφορά την ε, οικονομική ενίσχυση και την εκπαίδευση των γυναικών. Η συνάδελφός μου, κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, ε, ασχολείται ιδιαίτερως με τα ζητήματα αυτά ισότητα των φίλων και θέλει μέσω εφιών πολιτικών να βελτιώσει την κατάσταση, ιδίω στην Αφρική και σε άλλες περιοχές όπου οι γυναίκες ε, πλήττονται δυσανάλογα από την ε, ανέχεια και τα όσα αυτή συνεπάγεται. Στη Νέα Υόρκη ήρθαμε αντιμέτωποι και με την κατάσταση που ανέφερε η κυρία και Είχαμε δύσκολες συζητήσεις με τους αδέλφους από Πολωνία και Ουγγαρία και αυτό δεν είναι μυστικό για το πώς εμείς ε, θεωρούμε τα δικαιώματα αναπαραγωγικής ε, υγείας ε, των γυναικών. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και η προσέγγιση των Ούγγρων και Πολωνών συναδέλφων αντικατοπτρίστηκε και στην πρότασή μας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα διεκτησίας για τα ε, ζευγάρια, τα άγαμα μεν που όμως ε, έχουν συνάψει συμφώνω συμβίωσης. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, προτεραιότητες και κατευθύνσεις από τις επιμέρους κυβερνήσεις. Είναι διαφορετική προσέγγιση λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και ένας διαρκής διάλογος. να συζητήσουμε και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε ε, και τι μπορούμε να πετύχουμε. Δύσκολη νομίζω θα είναι και η συζήτηση για το σχέδιο δράσης ε, για τους ΛΟΑΔΜ και τη στρατηγική για το φύλλο στο επόμενο Συμβούλιο, γιατί αυτή είναι ακριβώς η χρονική στιγμή ε, που έρχονται στο προσκήνιο αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Ως προς τη μετανάστευση, Προσπαθούμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα από δύο οπτικές γωνίες. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το θέμα και στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και σε τα κέντρα και στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση γυναικών και εγώ και ο συνάδελφός μου κύριος Αβραμόπουλος που είναι επικεφαλής ε, ως προς τη διασφάλιση ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης, αλλά και των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά, την, ε, κατά τις διαδικασίες ε, που προβλέπονται από τη διαδικασία ασύλου, την πολιτική ασύλου. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε τις καλύτερε δυνατές ε, συνθήκε για τις γυναίκες και τα παιδιά και να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά ε, και στο ε, θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων. Βέβαια, ένα είναι ένα ευρωπαϊκό τέτοιο κείμενο και είναι κάτι διαφορετικό μετά πώς τα κράτη-μέλη θα μεριμνήσουν για τους μετανάστες και πώς θα εφαρμόσουν ένα κοινό τέτοιο κείμενο. σε ό,τι φορά την ε, παρακολούθηση είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι ε, συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων. Εξετάζουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε βασική ασφάλεια αντιμετώπισης του κινδύνου ε, μαστροπίας εμπορίας ανθρώπων, υποχρεωτικών εξαναγκαστικών γάμων και άλλων τέτοιων φαινομένων που απαντώνται σε χώρους ε, με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σοβαρό πρόβλημα φέτος. Θα υπάρξουν και άλλα βέβαια στην πορεία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όμως είδαμε πέρυσι 80% των μεταναστών ήταν νέοι άντρες. Φέτος η πλειονότητα των, γυναικών, ε, των μεταναστών είναι γυναίκες και παιδιά. Ιδίω ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Στη Σουηδία, στη Γερμανία, ανήλικοι που πέφτουν θύματα ε, επιθέσεων, αποσημωρίες. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε, αλλά και τα κάτι μέλη που βρίσκονται ε, στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή ε, και είναι αρμόδια για την προστασία αυτών των ατόμων. Μετά, κάτι το οποίο θα παραπευθεί και στο ζήτημα στο Συμβούλιο ε, Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν μετά οι μετανάστες την επόμενη μέρα, όταν εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Το συζήτησα με τους ε, ε, υπουργού δικαιοσύνη, ότι πρέπει να υπάρξει ένα στοχευμένο πρόγραμμα για τι γυναίκε ό,τι αφορά την εκμάθηση γλωσσών, ε, την προσφορά θέσεων απασχόλησης και τη διαμόρφωση ε, προϋποθέσεων για την παιδική μέρημνα. Και αυτό με φέρνει και στο ψηφιακό θεματολόγιο, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία να προσφέρουμε στις γυναίκες ε, διάβλους κοινωνικής ένταξης μέσω της ψηφιακής εποχής και των ψηφιακών δυνατοτήτων είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Αυτά για τη μετανάστευση. Πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη συστάση της κυρίας Χάνιμπολ και την έκθεσή της, γιατί εκεί αναφέρονται όλα όσα πρέπει και μπορούμε να κάνουμε. Όχι μόνο πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και πρώτα και κύρια από πλευράς κρατών μελών. Και η ενσωμάτωση των μεταναστών λοιπόν είναι κάτι που αναφέρεται ε, και στο θεματολόγιο δεξιοτήτων. Δεν ξέρω αν έχω άφησε κάτι. Έκθεση για την ενδυνάμωση των γυναικών ε, ε, στη ψηφιακή εποχή. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο θεματολόγιο δεξιοτήτων και αυτό μπορείτε να το ελέγξετε και πάλι, θα το δείτε ότι θα το εντάξουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιούροβα για την τόσο λεπτομερή εξειδικευμένη τοποθέτηση για πολλά από αυτά τα θέματα. Αληθεύει ότι πολλές φορές δεν έχουμε την απάντηση που θα μας, θα μας ευχαριστούσε. Διότι υπάρχει γενικευμένη εντύπωση, όπως εδώ αναφέρθηκε, ότι για συγκεκριμένα θέματα εξετάζοντας από την αρχή μια της κοινοβουλευτικής θητείας πολλές φορές ε, δεν υλοποιούνται λόγω τροχοπέδησης στο Συμβούλιο, άλλες φορές λόγω αποφάσεων που θεωρούμε ότι δεν ε, υιοθετούν και δεν προχωρούν ε, αυτά τα θέματα και αυτά όλα, ας το πω έτσι, απομένουν όσον αφορά τις πολιτικές και έχουν επιπτώσεις για τις πολιτικές ισότητας για τις γυναίκες. Αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας στο να εμείνουμε και να επιμείνουμε στην ανάγκη του να συνεχίσουν και να προαχθούν οι πρωτοβουλίες στο νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε άλλα επίπεδα όπως εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε. Ξεκινάμε τώρα το δεύτερο γύρο παρεμβάσεων ώστε να παρέμβουν οι ευρωβουλευτές ε, ατομικά τώρα στις παρεμβάσεις τους. Υπενθυμίζω ότι οι παρεμβάσεις θα είναι ενός λεπτού παρεμβάσεις για να μπορέσουν όλοι και όλες να παρέμβουν όσοι επιθυμούν, όσες επιθυμούν. κυρία Κοράτσα Μπίλτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, πραγματικά για το στένο και την εμπλοκή σας ε, για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φίλων Απαντήσατε πολλά από τα θέματα που με ανησυχούν και είναι μελήματά μου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την επικέντρωσή σας στην πρόληψη και καταπολέμηση βίας όσον αφορά την βία κατά των γυναικών. Και έγινε λόγος ήδη για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πραγματικά καλωσορίζω την επικέντρωση σε σχέση με αυτό. Θα είναι μια μακρά διαδικασία δυστυχώς, χρονοβόρα και μακρά. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο συνεκτικός τρόπος και αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της βίας. Ποια είναι Ποιε είναι οι συγκεκριμένε δράσει ε, για να ενθαρρυνθούν και να προτραπούν τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα για να κινητοποιηθούν και εκείνες, εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν επικυρώσει να υλοποιήσουν τελικά, να εφαρμόσουν αυτή τη σύμβαση για την έκθεση, για την ε, υλοποίηση της οδηγίας για το ανθρωποεμπόριο. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν έχουμε την έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέμα το οποίο είχαμε εξετάσει σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε, ποια είναι η πρόοδος και τι γίνεται σε σχέση με τις δράσεις, μια και η ανθρωποεμπορία δυστυχώς εμπλέκει όλο και περισσότερες γυναίκες και παιδιά και είναι πραγματικά συντριπτικά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τη μετανάστευση για αυτό το θέμα. Το τρίτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ήθελα να μου αρέσει η έκφραση Team Europe, η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Σύνοδο Κορυφή στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω ότι το ίδιο θα μπορέσει να γίνει και για την Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχει το έργο με τους συναδέλφους σας επιτρόπους για να καταλήξετε στις πολιτικές αυτές για την ισότητα, στις συνολικές πολιτικές για τα θέματα των κοριτσιών όσον αφορά τον ακροτηριασμό, γενετή, το, γενετήσιο ακροτηριασμό ε, γυναικών, ε, κοριτσιών και θέματα τα οποία έχουν ήδη και προαναφερθεί και τα θέματα που αφορούν την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των κοριτσιών και γυναικών στις δράσεις μας. Στη Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη ελπίζουμε ότι θα ενταθούν αυτά και θα εξεταστούν και θα προέρχονται από μια φωνή που θα αρθρώνει λόγο συνεκτικό, ενωμένο από πλευρά της Ευρώπης, αποτελεσματικό για το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξή. Μια και κάνουμε λόγο για την προσχώρηση. Βρίσκεται καθοδόν αυτό, είναι υπό σε σχέση με το θεματολόγιο σας για να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα θέματα των δικαιωμάτων και των παιδιών. Ευχαριστώ. Και ε, ε, ε, ευχαριστώ και που μου δώσατε και μέρος του, από τον χρόνο σας από πλευρά συναδέλφου. Εσείς συνάδελφοι έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να προσθέσω τη φωνή μου στους επένους που ακούστηκαν. Θέλω επίσης να εκφράσω και την εξή τοποθέτηση. Είμαι ανυπόμονη και η ανυπομονησία ανήκει στο κίνημα των γυναικών. Επί ε, αιώνες αναμένουμε για την ισότητα και ανυπομονώ ακούγοντας πόσο μικρά βήματα γίνονται για να σημειωθεί πρόοδος. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω και θα ήθελα να μου δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Κυρία Επίτροπε, για την ερώτηση ποιες δυνατότητες υπάρχουν την ε, ενσωμάτωση επαγγελματικά των γυναικών για τις γυναίκες και για τις τυπικές επαγγελματικές ε, εργασίες των γυναικών. Θα ήθελα επιτέλους να μπορέσουν να πληρωθούν ε, όπως θα έπρεπε. Αν <clears throat> πραγματικά πληρωνόντουσαν όπως θα έπρεπε θα υπήρχε ανταγωνισμός για να καλυφθούν αυτές οι εργασίες, αυτές οι δραστηριότητες και από άντρες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Μία ερώτηση έχω. Είπατε στα όσα εκθέσατε με σαφήνεια ότι τα κράτη-μέλη με, με νομική δράση προχώρησαν και πάντα τότε υπήρχαν επι, επιτυχίες λέτε. Δεν γίνεται λοιπόν με παρακλήσεις με το να παρακαλάμε και τα παρακάλια. Πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική στεναρή δράση. Σας ερωτώ λοιπόν, τι κάνετε εσείς Επίτροπε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα, ώστε τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν, να μην καταλήγουμε σε μια κατάσταση με παρακάλια, παρακαλώ, παρακαλώ βοηθήστε, αλλά νομικά βήματα και διαβήματα να αναλυθούν υπέρ της ισότητας. Ευχαριστώ. Σεμπαστιά, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, κυρία Γιουρόβα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και να έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Εγώ ως μέλος πρέπει να πω ότι είχα ξεχάσει σε σχέση με τη, τους επιτρόπους ε, τα χαρακτηριστικά τους. Με σας δεν συμβαίνει αυτό γιατί προσέρχεστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, δεν θα κατονομάσω, αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο αφορά το, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υιοθετήσει, να προσχωρήσει στην σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Φοβούμαι ότι είναι τα ίδια που μας είπατε και στην τελευταία μας συνάντηση, στη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο. Τότε ήταν χειμώνα, δεν ήταν άνοιξη όπω τώρα. Πέρασε χρόνο από τότε. Διαρωτώ με, μπορείτε να μα δώσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για αυτή την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζω ότι μόνο τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα κατά τη βία ή ανισότητα κατά των γυναικών. Αλλά το πολιτικό μήνυμα είναι ισχυρό. Πρέπει να αποσταλεί στα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα. Λοιπόν, το δεύτερο αφορά την βία με βάση το φύλλο. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Αλλά γνωρίζουμε δεν είναι άποψή μας, το διαβάζουμε και στις απόψεις ε, του Ιδρύματος, Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Ισότητα και τις ε, υπηρεσίες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι κάποιες προσπάθειες είναι ιδιαίτερα αποδυναμωμένες και όχι αποτελεσματικές. Έχουμε σημαντικό πρόβλημα εδώ. Δεν έχουμε το κοινό εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει, ας το πω έτσι, ε, η νομική, νομοθετική δυνατότητα ώστε σε νομοθετικές κατηγορίες, για παράδειγμα πραγμάτων, ε, εγκλημάτων που αποκαλούμε ε, εγκλήματα ε, που το πάθος οδήγησε σε κάποιους να εγκληματίσουν. Θα πρέπει να είμαστε πιο εξειδικευμένοι. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες εξειδίκευσης και ανάληψης πρωτοβουλειών. Μπορείτε να βασίζεστε σε μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεμπαστιά. Η κυρία Σόντροβα τώρα θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την πολύ πρακτική προσέγγιση, χειροπιαστή προσέγγιση σε αυτό, το θεματολόγιο. Επανειλημμένα ανέφερε ότι η ίδια η νομοθεσία αυτής δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε την εφαρμογή, στην πρακτική καθημερινή εφαρμογή των μέτρων αυτών που συζητούμε και διαβουλευόμαστε επ' αυτών. Συνάδελφοι, Γνωρίζουμε ότι η αρνητική μεταχείριση με βάση το φύλλο απαγορεύεται και όμως παρόλα αυτά υπάρχει και το μισθολογικό χάσμα. Οι διαφορές δηλαδή μεταξύ μισθών γυναικών και ανδρών. Υφίστανται αυτές οι διαφορές και η άνηση αυτή ε, πληρωμή των γυναικών και έχουμε αυτή την κατάσταση όχι μόνο στους μισθούς. Απαγορεύεται η αντική μεταχείριση και όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πηγές μη νομοθετικού χαρακτήρα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή και τα πράγματα χωλένουν. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν κάτι επιτέλους για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε λοιπόν, να, ληφθεί, να σας ζητήσω να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάποιας έρευνας για τη συνεισφορά στο, στον τομέα αυτό. Γυναικών δηλαδή που, που εμπλέκονται και συμμετέχουν στην περίθαλψη και φροντίδα παιδιών και εκείνων που δεν το κάνουν. Γονείς ε, οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά τους πραγματικά όσον αφορά το εισόδημά τους υφίστανται αρνητική μεταχείριση. Αν μπορούμε έτσι να τεκμηριώσουμε τα πράγματα θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε τις λύσεις που είναι αναγκαίες για τους γονείς που φροντίζουν τα παιδιά. Αν μια μάνα μένει στο σπίτι και έχει ένα παιδί που φροντίζει, μετά ακολουθεί ένα δεύτερο παιδί, μετά από τρία-τέσσερα χρόνια μια τέτοια γυναίκα ξεκινά από μια τελείως διαφορετική αφετηρία την επαγγελματική τη ζωή ή τη συνεχίζει από τελείως διαφορετική αφετηρία. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί. Για την πρόταση στο έγγραφο εργασίας ότι 40% των εργαζόμενων γυναικών που σε υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να, συμμετέχουν. Θα ήθελα να μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα και διαβήματα. Ποια είναι αυτά τα εξειδικευμένα βήματα. Είναι ο καλύτερος τρόπος από ό,τι νομίζω για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο η κυρία Δάντσιλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως με την προσέγγισή σας, διότι τα θέματα τα οποία φύγετε ε, είναι θέματα τα οποία μας ανησυχούν, μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή μας αλλά αποτελούν και θέματα τα οποία απασχολούν κάθε κράτος μέλος. Είπατε ότι το 2017 θα είναι το έτος ε, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένος μέσω ψηφισμάτων του έχει ζητήσει την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την ε, ε, βία ε, λόγω φύλου για, ως τμήμα του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια ώστε να μπορέσει το Ινστιτούτο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ποια είναι η απόψή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και για να ολοκληρώσουμε με τις παρεμβάσεις, η κυρία Ροντρίγες. Ευχαριστώ για την παρουσία σας κυρία Πίτροπε και συγχαίρω για τις προσπάθειες που έχετε κάνει σε σχέση με το, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ερωτήσεις μου αφορούν τα εξή Σε σχέση με τη μετανάστευση και για τα θέματα ασφάλειας όσον αφορά τις γυναίκες και το, τους LGBT από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται, ποιε είναι οι κυρώσει ε, για τι χώρε εκείνε που δεν υλοποιούν ε, τι προδιαγραφέ για τι γυναίκε και ε, του LGBT. Και ένα άλλο θέμα σε σχέση με το ΕΛΚ. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η καταπολέμηση του γενετήσιου ακροτηριασμού των κοριτσιών σε σχέση με τα στοιχεία δεν ήταν σαφή όσον αφορά την, ε, ε, τον έλεγχό τους και την επαλήθευσή τους. Και στο τέλος μια πιο προσωπική ερώτηση για την πολιτική αποσαφήνιση. Θα ήθελα να ξέρω κυρία Επίτροπε για την κατάσταση της Air France που υποχρεώνει τις υπαλλήλους ε, να καλύπτουν το πρόσωπό τους στις πτήσεις στο Ιράν. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος αρνητικής μεταχείρισης αυτών των υπαλλήλων της Air France. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις ε, και τα σχόλια των ε, Ευρωβουλευτών. Καταρχάς, στην κυρία Κοράτσα η οποία ρώτησε και αναφέρθηκε και πάλι στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πώς ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη. Ε, πιέζουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε μόνο. Χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία. Όπως σας είπα για μένα, η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν θα μπορέσει να βοηθήσει να υλοποιηθούν όλα τα καθήκοντα από πλευράς κρατών μελών, κυρίως όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη, χωρίς να υπάρξει κατάλληλη ε, συμπερίληψη των ε, αδικημάτων αυτών στην νομοθεσία. Δεν θα υπάρχει ποτέ κάποιος ανασταλτικός παράγων για τους εγκληματίες. Επομένως, ε, αυτό πρέπει να το επιτύχουμε. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο νομοθετικό μέσο για να τους πιέσω να κυρώσουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόσκομα από πλευράς κατών μελών. Ένα γενικό σχόλιο τώρα για να απαντήσω και σε κάποια από τα σχόλιά σας ε, που ε, ζητούν νομοθεσία. Βεβαίω και η νομοθεσία είναι το ιδανικό μέσο όταν πρέπει να πιέσουμε κάποιον να κάνει κάτι ή να αποθαρρύνουμε κάποιον μέσω νομικών μέσων. Ε, ε, να τον αποτρέψουμε από το να κάνει κάτι. Αλλά το ξέρετε κι εσείς ότι τα θέματα φύλου συνδέονται πολύ και με παραδόσεις και με στερεότυπα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν απλώς ε, με νέα νομοθεσία. Και κάτι το οποίο συνειδητοποίησα 1,5 χρόνο ε, όντας εδώ, όταν ε, ε, μια νέα νομοθεσία απλώς ε, της δώσουμε ένα τίτλο που αναφέρεται στο φύλλο δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν λειτουργεί αποτελεσματικά σίγουρα στους κύκλους μας και σε καμία περίπτωση δεν έχει αποτελέσματα σε κάποια κράτη-μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη για να είμαι πιο συγκεκριμένη. Γι' αυτό και για να υπάρχει για το θέμα της ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου προσπαθώ να εξηγήσω όταν μιλάω σε διάφορα βήματα τις οικονομικές συνέπειες θετικές ε, συνέπειες ε, της άρσης ε, των φραγμών για γυναίκες που έχουν παιδιά και να μπορούν ταυτόχρονα και να εργάζονται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα με την νομοθεσία και το δεύτερο είναι ότι συνήθως όταν έχουμε νομοθεσία η οποία η οποία έχει και συνέπειες για τον προϋπολογισμό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι το θέμα με την οδηγία κατά των διακρίσεων, την οποία προωθούμε και ξέρετε ότι χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο και ακόμα αρκετά κράτη-μέλη δεν ε, συμφωνούν. Και το βασικό του επιχείρημα μεταξύ άλλων είναι ότι δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αυτά είναι γενικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν με την ομοθεσία. Όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, η Επιτροπή παρακολουθεί την μεταφορά της οδηγίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων. Τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να μεταφέρουν ε, την οδηγία μέχρι τον Απρίλιο του 2013. 26 κράτη-μέλη μέχρι σήμερα έχουν ενημερώσει επισήμω ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει γίνει μεταφορά τη οδηγία σε εθνικό επίπεδο και υπάρχει ενημέρωση ότι πλέον επετέχθηκε η πολιτική συμφωνία και στη Γερμανία. Περιμένουμε λοιπόν και τη σχετική επίσημη κοινοποίηση. Άρα, 26 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύονται από την ε, οδηγία έχουν κοινοποίησει πλήρη μεταφορά. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου Βραμόπουλου και οι υπηρεσίες του αυτή τη στιγμή αναλύουν τις πληροφορίες ε, οι οποίες κοινοποιήθηκαν επισήμως από τα κράτη-μέλη. Για το Team Europe, αυτή την ε, ομαδική δράση από πλευρά Ευρώπη, το ένιωσα και εγώ στη Νέα Υόρκη και ήταν σημαντικό όχι μόνο το γεγονό ότι συναντηθήκαμε εμεί, γιατί όπω σα είπα υπήρχαν αρκετέ σημαντικέ συνεδριάσει, αλλά το γεγονό ότι ε, συναντήσαμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Και επειδή δεν υπάρχει πρόοδος ε, στα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα, διαπιστώνω ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί καλό παράδειγμα για τις γυναίκες. Και όσον αφορά και κάποιες ερωτήσεις σας για την καλύτερη ισορροπία και το, διαφορά μισθών, να σας πω ε, άκουσα ένα σχόλιο ότι τα μοντέλα ε, δουλεύουν δωρεάν. Οι μητέρε, δουλεύουν δωρεάν, συγγνώμη. Σχεδιάζουμε κάποια πράγματα προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκε εργασία για εργαζόμενους γονείς. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα, οι γυναίκε να πληρώνονται ε, για τον κόπο τους, για το ό,τι κάνουν στο σπίτι, να το εκτιμά αυτό η κοινωνία. Και ε, άρχισε να γελάει ο συνομιλητέ μου και νόμιζε ότι αστείευομαι. Τι, θα πρέπει να πληρώνονται για τις ε, για τα οικιακά τους καθήκοντα, ναι, τους είπα, γιατί το χρειάζεται η κοινωνία αυτό που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι, χρειάζεται τη δουλειά τους και κατάλαβα ότι είναι με πολύ διαφορετικός ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και ε, αυτό ε, δεν απέχει πολύ από τις συζητήσεις που κάνω με κάποιους Ευρωπαίους πολιτικές, πολιτικούς για να καταλάβετε λίγο και πού βρισκόμαστε. Τώρα, ε, ε, κάποιες ε, διακρίσεις και, κλειστά επαγγέλματα. Έχω πρόβλημα. Πρέπει να συναντηθώ με συνδικάτα που θα πρέπει να πιέσουν ώστε ε, να είναι πιο ανοιχτά κάποια επαγγέλματα. Σίγουρα πρέπει να το αυξήσουμε αυτό και πρέπει να σας πω ότι είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας επιβολή κυρώσεων στα κράτη-μέλη σε περίπτωση διακρίσεων και αυτό θα το κάνουμε. Αλλά αυτό είναι μόνο τμήμα του προβλήματος, το γεγονός ότι οι άνδρες πληρώνονται ε, για την ίδια δουλειά περισσότερο από ότι μια γυναίκα. Ε, η, ε, τα επαγγέλματα αυτά τα οποία δεν είναι ανοιχτά προς το ένα το άλλο φύλλο είναι το πρόβλημα. Το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν και πώς μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι στον τομέα αυτό είναι σημαντικό. το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Σα είπα ότι κάθε φορά που έρχομαι και σα λέω τι ίδιε πληροφορίε, ε, ε, ανησυχώ. Δεν είναι απόλυτα σωστό βέβαια αυτό για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχει υπάρξει πρόοδος, ε, θέλαμε να τελειώσει μέχρι φέτος. Υπάρχουν συζητήσεις τώρα στο Συμβούλιο και να σας πω ότι τα κράτη-μέλη που στηρίζουν την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη και απλώς ευκρινίζουμε κάποιες λεπτομέρειες τώρα, κυρίως ε, ποιες είναι οι ανησυχίες των κρατών μελών, ποια είναι η νομική βάση και ποιες θα είναι οι νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της προσχώρησης στη Σύμβαση. Και περιμένουμε φυσικά και την απόφαση του Συμβουλίου για το χειμώνα φέτος. Ο χειμώνα βέβαια μπορεί να σημαίνει 2016 αλλά και 2017. Ελπίζω να είναι φέτος για την ε, προσχώρηση της σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, ε, δεν σκοπεύουμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ποιος ρώτησε. Περισσότερες γυναίκες στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 40% είναι γυναίκες. Νομίζω ότι πολύ σωστά ε, αντικατοπτρίζεται αυτό στο νέο ε, γύρο για νέους διευθυντές γενικών διευθύνσεων και αυτό δεν ήταν μόνο η δική μου η προσπάθεια για να υπάρχει εξορθολογισμός, αλλά πρέπει να σας πω ότι και η Κρυσταλίνα Γεωργίευα ε, είναι αφοσιωμένη στο στόχο αυτό των περισσότερων γυναικών και προωθεί συγκεκριμένες γυναίκες σε συγκεκριμένες διευθυντικές θέσεις και λέει ότι είναι εξαιρετική γυναίκα πάντα. Και μ' αρέσει να την ακούω να το λέει αυτό γιατί συνήθως έχει δίκιο. Το 40% μπορεί να επιτευχθεί αλλά χρειάζεται μόνιμη πίεση από όλου ε, τους ευθύνοντες και φυσικά να υπάρχουν και γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα του συστήματος γυναίκες στην πρώτη γραμμή. Αυτά σας ευχαριστώ. Thank you, ε, ευχαριστώ κυρία Γιούροβα. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην ε, συζήτηση αυτή, στην ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμικό τρόπο και μακάρι την επόμενη φορά που θα έρθετε εδώ στην Επιτροπή μας να υπάρχουν θέματα στα οποία αναφερθήκαμε σήμερα, τα οποία να μπορούμε να τα έχουμε μεταφράσει σε συγκεκριμένες πράξεις. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης Προϋπολογισμός 2017. Ε, Συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Ντανσίλα, στην οποία δίνουμε και το λόγο για να μας παρουσιάσει το περιεχόμενο της γνωμοδότησής της. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης για το σχέδιο προπολογισμού 2017 ω προς την Επιτροπή Γυναικών έχουμε αναφέρει τι προτεραιότητε ε, της Επιτροπής μας σε διάφορους ε, τομεί πολιτική, Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη συνεκτική αξιοποίηση του προπολογισμού για την ισότητα μεταξύ των φύλων σε όλα τα στάδια της ε, διαδικασία προπολογισμού. Δεύτερον, χρήση των διαφορετικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων για την προώθηση της ε, ποιοτική εκπαίδευσης, της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά και της δημιουργίας ε, ε, θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες. Τρίτο σημείο προτεραιότητες, επαρκή πόροι για το πρόγραμμα Δάφνη, ειδικέ δράσεις και κονδύλια για τις μετανάστριες και, τους, και τις γυναίκες του άσυλο και τέταρτον ισότητα των φύλων, όπως και ανέφερα στην Επίτροπο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ζητήσει σε ψηφίσματά του τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ισότητα μεταξύ των φίλων Αυτά είναι τα πέντε σημεία που αποτελούν προτεραιότητε βάσει και τη δική μου έκθεση. Περιμένω να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων. και θα πρέπει να τηρηθεί και η προθεσμία. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΚ, κυρία Κονόσκα, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαδέρα δεν είναι εδώ. Ζητεί συγγνώμη. Μου άφησε ορισμένες σημειώσεις και θα θέλω να τις διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νταντσίλα για το έργο της. Έχουμε παρατηρήσει ότι συμπεριλαμβάνει στην γνωμοδότηση πολλά από τα αιτήματα που κάναμε από πλευράς ΕΛΚ πέρσι, όταν το ΕΛΚ ήταν, ε, είχε αναλάβει αυτή την γνωμοδότηση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία χρηματοδότηση των μέτρων που έχουν ως στόχο τη στήριξη τη ποιοτική ε, εκπαίδευση, τη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ως ΕΛΚ στηρίζουμε πλήρως αυτό που αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού για τον Δάφνη. Και βλέπουμε ότι και οι σοσιαλιστές συμφωνούν μαζί μας. Αντί να δημιουργήσουμε ένα νέο οργανισμό συγκεκριμένα για τη βία κατά των γενικών, θα ήταν πιο χρήσιμο να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, για την ισότητα μεταξύ των φίλων και να έχει νέο προσωπικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντκε παρακαλώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της συναδέφου Μόνικα που βρίσκεται σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Θα αναφέρω κάποια σημεία που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά για αυτό το ζήτημα. Για την νομοδότηση δηλαδή. Το πρώτο σημείο. Το χαιρετίζουμε ιδιαίτερα ότι στον προϋπολογισμό, στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, αυτό θα διαδραματίζει ένα κέριο ρόλο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επικοδομητικό μέτρο ώστε ο προϋπολογισμός να γίνει πιο δίκαιος όσον αφορά τη διάσταση του φύλου. Και από πλευράς της εισηγήτριας θέλουμε να ευχαριστήσουμε ότι τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο στο σχέδιο αυτό. Το δεύτερο σημείο το οποίο χαιρετίζουμε ιδιαίτερα είναι σε σχέση με την νομοθεσία τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ε, έχουμε θέσει κέντρα βάρους και ένα από τα κυριότερα θέματα των επόμενων μηνών θα είναι ακριβώς να αναφερθούν τα θέματα αυτά που θα πρέπει να εντάσσονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ένας, ε, μια κύρια ομάδα που θα αφορά και την χρηματοδοτική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί είναι θετικό ότι με κέριο ρόλο αυτό εντάσσεται σε αυτή τη γνωμοδότηση. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο η συνάδελφος θα ήθελε να τονιστεί ιδιαίτερα, είναι το θέμα του πώς θα έχουμε μια θετική πρόσβαση για τις γυναίκες, για το, το επάγγελμα που ασκούν, για τη σταδιοδρομία τους, όχι μόνο σε σχέση με τις, το ρόλο τους ως καταναλωτών, αλλά για την απασχόληση Όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες που παρέχονται, θέλουμε ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη τα θέματα των γυναικών και να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια για το έργο που έχει επιτελέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς και για να ολοκληρώσουμε το γύρο των παρεμβάσεων. Εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Yes, and, ε, Ευχαριστώ. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω λέει η κυρία Μούντι την εισηγήτρια για το ρόλο που έχει διαδραματίσει. Είναι πολύ θετικός και χαιρετίζουμε την διάσταση του φίλου στα θέματα προϋπολογισμού και στην αντιμετώπιση θεμάτων όσον αφορά διαφορές που υφίστανται σε σχέση με τις, ε, το, τη διάσταση του φύλου εις βάρος των γυναικών, ώστε κορίτσια και γυναίκες να μπορέσουν να λυθούν ιδιαίτερα και γυναίκες ετούντες άσυλο, ετούσες άσυλο επίσης τελευταίο που θα ήθελα να πω, αντιμετωπίζοντας ε, την διαμόρφωση του φύλου στα, στον προϋπολογισμό πρέπει να έχουμε μετρήσιμους στόχους και να δούμε το πώς αυτοί οι στόχοι θα μπορέσουν να δώσουν ένα feedback ε, για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε δράσεις που έχουν αποτέλεσμα και αντίκρισμα. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο, η κυρία Ντανσίλα θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, η κυρία Ντανσίλα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ τις συναδέλφους που υποστηρίζουν τα θέματα στην έκθεση και τις προτάσεις ε, τους. Σίγουρα όταν θα έχουμε τις τροπολογίες ε, θα έχουμε πλέον ένα σχέδιο γνωμοδότησης που θα αντανακλά ε, την ίδια την πραγματικότητα και έτσι θα εστιαστούμε στα θέματα των γυναικών στον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα που έχει εγκριθεί. Στις 28 Απριλίου ολοκληρώνεται η κατάθεση τροπολογιών. 24 Μαΐου θα εξεταστούν αυτές οι τροπολογίες. 13-14 Ιουνίου ψηφίζουμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, 30 Ιουνίου στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προϋπολογισμών και τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Και περνάμε στο τελευταίο μα σημείο στην ημερησία διάταξη που είναι η έκθεση για την προετοιμασία της αναθεώρησης όσον αφορά τις δημοσιονομικες δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2017. Κυρία Μούντιν, θα έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δεν θα είναι μεγάλη έκπληξη, αλλά και εδώ έχουμε πάλι το gender budgeting, θέμα δηλαδή διαμόρφωσης θεμάτων χρηματοοικονομικών και κονδυλίων από πλευράς προϋπολογισμού για την ισότητα. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τον προϋπολογισμό σε ένα μακρότερο επίπεδο χρονο, ε, ε, χρονικό και όχι μόνο ετήσια. Αντανακλώνται λοιπόν αυτά, αυτές οι ανάγκες. Ε, στρεφόμενοι στους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, βλέπουμε ότι αυτά όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2017 αυξάνοντας την απασχόληση για τις γυναίκες πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το αίτημα για τους ίσους μισθούς, την ίση ανταμοιβή για ίδια εργασία και σε σχέση με την μέτρηση πώς αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται. Επίσης με κοινή δήλωση για το gender mainstreaming, την ενσωμάτωση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Χρειαζόμαστε δράσεις για το follow-up, για την παρακολούθηση και συνέχεια που θα δοθεί περισσότερα να γίνουν για την υλοποίηση και εφαρμογή και όχι μόνο ωραία και καλά λόγια και ένα περιεχομένου. Και εδώ πάλι το θέμα το οποίο αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση για την βοήθεια την οποία πρέπει να προσφέρουμε στις γυναίκες ετούσες άσυλο, γυναίκες πρόσφυγες και γυναίκες μετανάστριες και με την ενίσχυση κονδυλίων και επενδύοντας στις κοινωνικές υποδομές χρησιμοποιούμε μια διαφορετική προσέγγιση για το τι σημαίνουν οι υποδομές ε, σε σχέση με τις δράσεις μας. Να μπορέσουμε τις γυναίκες δηλαδή να τις περάσουμε και στην απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η προσέγγιση και η άποψή μας όσον αφορά τις δράσεις και τις υποδομές. Και τέλος να διασφαλίζεται και η διαφάνεια του προγράμματος Δάφνη να είμαστε σε θέση να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε αυτό που είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα κατά της βίας κατά των γυναικών, του προγράμματος Δάφνη δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μούντι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να ζητά τον λόγο να παρέμβει, πράγμα που σημαίνει ότι οι βουλευτίνες που βρισκόμαστε εδώ συμφωνούμε απόλυτα με την παρουσίαση που έγινε από πλευρά σας. Και έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής για σήμερα, ευχαριστώντας για την υπομονή σας και ελπίζω να σας ξαναδούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Γεια σας.